Präsident! Guten Meine αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση που στις 13 Δεκεμβρίου του 2012 διεκόπη, συνεχίζεται με σημερινή ολομέλεια.